Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ ας ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε ένα επιφανή καλεσμένο σήμερα το πρωί και φαντάζομαι πολλοί συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο αργότερα στη συζήτηση. Συζήτηση που θα ξεκινήσει όσον ούπο. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Ως συνήθως ε, μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής. Πριν περάσουμε στο διάλογο το διαρθρωμένο με τον Επίτροπο Τιερή Μπρετό θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση γιατί είναι η τελευταία φορά που έχουμε μαζί μας συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Επιτροπή. Θα ήθελα εκ μέρους ε, και μου και της Επιτροπής και της ε, Γραμματείας να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Επιτροπής μας από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ανεκτήμητη συμβολή τους. Λυπάμαι που το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σεβαστούμε τη βούληση του Βρετανικού λαού. Και προσβλέπουμε σε μια νέα καλή σχέση με, την, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο που θα εδράζεται στις ίδιες ε, αξίες και αρχές και ενδιαφέροντα που μοιραζόμαστε και που είναι πολλά. Ελπίζω ότι η νέα μας σχέση θα είναι ισχυρή ιδιαίτερα για το πλαίσιο ορίζων και για την έρευνα, αλλά και για πολλά άλλα θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν την Επιτροπή και ενδιαφέρουν φυσικά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία και με το νέο πλαίσιο των σχέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο και να τους αποχαιρετήσω. Και να καλωσορίσω ταυτόχρονα τον Επίτροπο Τιερή Μπρετών, τον Επίτροπο εσωτερική αγορά, όπω ξέρετε, που έχει όμω ευρύτερο το χαρτοφυλάκιο, την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, μικρομεσαίε επιχειρήσει, διαστημική πολιτική και ψηφιακή πολιτική. Και τον ευχαριστώ θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε εδώ ε, τον ε, Επίτροπο μετά την ανάληψη των ε, καθηκόντων του, τον είχαμε στην ακρόαση της επιβεβαίωσης, θα θέλαμε να ακούσουμε τι γίνεται με την βιομηχανική πρωτοβουλία και την πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναμένεται για το Μάρτιο και για πολλά θέματα, για την αμυντική μας βιομηχανία, τι θέση θα έχει στη βιομηχανική πολιτική και επίση ε, ποιο είναι το επικείμενο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα που σχολιάσαμε και με άλλου συναδέλφου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Επίση για τα δεδομένα. Ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλέ στον Επίτροπο ε, και για το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρουσε ιδέε. Επίση ε, θα έχουμε αρκετά κονδύλια για το νέο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Ε, στην, ε, στις διαπραγματεύσεις ε, της επικείμενες για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Ένα τέταρτο θα μας μιλήσει αρχικά ο Επίτροπος. Θα ακολουθήσει ο πρώτος γύρος των ρωτοπαντήσεων με τους συντονιστές και θα έχουμε και δεύτερο γύρο με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Εκεί όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούσα να λάβουν το λόγο. Και Όταν θα ξεκινήσει την ομιλία του ο Επίτροπος, ήδη δηλώστε ποιοι θέλετε να λάβετε το λόγο στη συζήτηση. Σηκώνετε την καρτέλα σας και αφήνετε την όρθια για λίγα λεπτά, προκειμένου να σας καταγράψει η γραμματεία και να μην ξεχάσει κανέναν. Βλέπω μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Ήδη έχουμε σίγουρα 20 ομιλητές στον κατάλογο και δεν έχει καν ξεκινήσει ο Επίτροπος την ομιλία του. Αφήστε λοιπόν το καρτελάκι σας ε, όρθιο για να σας σημειώσει η γραμματεία. Και τώρα να καλέσω τον Επίτροπο Μπρετόν που για ένα τέταρτο θα μας εξηγήσει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το όραμά του για τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Και αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν τα γαλλικά μπορούν να με ακούσουν από τη διερμηνία. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, κύριε, κυρίες και κύριοι της ε, Επιτροπής, είναι μεγάλη τιμή για μένα που για πρώτη φορά λαμβάνω το λόγο εδώ στην Επιτροπή σας. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε την ακρόαση και από την τελευταία μας συνάντηση έγινε σημαντική δουλειά για πολλά σημαντικά θέματα. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο τέταρτο που μου δώσατε, άντε 16 λεπτά, αλλά έχω τόσο ευρύ χαρτοφυλάκιο. Βιομηχανία, μικρομέσες επιχειρήσεις, διάστημα, άμυνα και την ψηφιακή Ευρώπη. Ένα ευρύτατο φάσμα λοιπόν θεμάτων. Και το πρόγραμμα μου είναι πολύ φιλόδοξο. Πολλές πρωτοβουλίες θα υποβάλουμε και μάλιστα και με άλλους συναδέλφους είχα επιτρόπους συζητήσει και με εσά, πολύ επικοδομητικές. Και σίγουρα όλες αυτές οι συζητήσεις ε, με βοηθούν για να διαμορφώσω αυτό το όραμα. 19 Φεβρουαρίου, σημειώστε τις ημερομηνίε για να τις έχετε κατά νου και να συντονιστούμε. 19 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσουμε τις φιλοδοξίες μας για τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αρχίζουμε και αγκύπτουμε στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης πιο διεξοδικά και θα διαμορφώσουμε και μια στρατηγική για τα δεδομένα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι απόρρια της στρατηγικής για τα δεδομένα. Γι' αυτό θα καλό είναι να έχουμε παράλληλες στρατηγικές και για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα και η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μου ανέθεσε και αυτό το έργο. Επίσης, 4 Μαρτίου θα υποβάλουμε την ε, βιομηχανική μας στρατηγική, όπως είπατε κι εσείς. Το έχουμε συζητήσει ήδη. Ε, θα σας παρουσιάσω τους άξονες του μετασχηματισμού, ψηφιακό, εμ, κρίσιμες τεχνολογίες ε, για να εξασφαλίσουμε την βιομηχανική μας κυριαρχία. Είναι θέματα και εσωτερικής αγοράς. Αύριο θα σας παρουσιάσουμε την ε, συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την θωράκιση των κρίσιμων δικτύων, πέμπτης γενιάς κυρίως, που είναι κρίσιμες υποδομές και ιδιαίτερα για τις βιομηχανικές εφαρμογές, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για μας και αφορά φυσικά το χαρτοφυλάκιό μου, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περιμένουμε ανυπομονησία τη συζήτηση μαζί σας για να συντονιστούμε και να διαμορφώσουμε από κοινό αυτή τη στρατηγική. Τώρα θα αγγίψω στην επιμέρους σημεία της στρατηγικής, ξεκινώντας από αυτά που είναι τα πιο σημαντικά. Καταρχήν ψηφιακό πακέτο, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Γενικώ. Όλοι συμμετείχατε με τον ΑΒ τρόπο στην ακρόαση πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, οπότε ξέρετε τα θέματα που γνωρίζω. Εγώ δεν συμφωνώ ότι στερούμε στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά και τα δεδομένα. Δεν θα πρέπει να δίνουμε αρνητικά μηνύματα. Σε, κάποια, σε κάποιους τομείς στερούμε, σε άλλα όμως προηγούμαστε. Αλλά τίποτα δεν έχει λήξει σε θέματα δεδομένων και κυρίως βιομηχανικών δεδομένων. Και θα επανέλθω στα θέματα αυτά. Φιλοδοξία της στρατηγικής μας είναι να απελευθερώσουμε αυτά τα βιομηχανικά δεδομένα. Και αν δούμε τι συνέβη με την δημιουργία των μεγάλων πλατφορμών, το πρώτο κύμα ήταν τα δεδομένα τα προσωπικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Και ο έλεγχος αυτού του τεράστιου όγκου των προσωπικών δεδομένων που γίνονται στην ε, Αμερική, στην Κίνα, γιατί εκεί υπάρχουν ολοκληρωμένες αγορές και ισχυρές αγορές δεδομένων. Μετά είχαμε κάποιες πρακτικές ε, απόκτηση, αγοράς δεδομένων και μάλιστα ε, είναι αμφισβητήσιμες μερικές φορές και προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποιες παρεκκλήσεις ε, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων. Πάντως, τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικοί παράγοντες εποφελήθηκαν από αυτή την συγκέντρωση δεδομένων για να προτείνουν κάποιες υπηρεσίες για προσωπική κυρίως χρήση. Πολύ συχνά αναφέρω ότι τα δεδομένα είναι τμήμα μιας κληρονομιάς. Προσωπικής κληρονομιάς και βιομηχανικής κληρονομιάς και επιχειρηματικής κληρονομιάς. Και τα δεδομένα που δημιουργούν οι επιχειρήσεις δημιουργούν νέες εμπειρίες και ε, δημιουργούν αλγορίθμους για νέες εφαρμογές. Οπότε, εδώ δεν μιλούμε για τεχνικά θέματα μόνο. Ε, η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων θα είναι ένα μεγάλο τμήμα του ε, ΑΕΠ, 700 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, διόλου καταφρόνει τη συμμετοχή και ποσό. Το καλό μαντάτο είναι, ε, και θα χρησιμοποιήσω εδώ ένα παραλληλισμό, σήμερα ο πλανήτης μας είναι 40 τετρά, εκατομμύρια και παραπάνω δεδομένα. Αυτή είναι η κληρονομιά των δεδομένων που δημιουργήθηκε από την αρχή των δεδομένων. Τόσα δεδομένα έχουμε αποθηκευμένα ε, που κάθε 18 μήνες ανανεώνονται και πολλαπλασιάζονται. Τώρα έχουμε 35 με 40 τετραμπάιτ και θα είμαστε σε 180 περίπου τετραμπάιτ πολλά, δισ, πολλά δισεκατομμύρια, Τρει τετράκι, πεντάκι εκατομμύρια δεδομένων. Τεραμπάιτ, 185. Οπότε ένα μεγάλο τμήμα τη παγκόσμια παγκόσμιας και ένα μεγάλο τμήμα ε, θα είναι στην, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στο μέλλον θα είναι αυτό που έχουμε σήμερα στο σύνολο του πλανήτη. Οπότε αυτό ενδιαφέρει κυρίως στις επιχειρήσεις, τα συνδεδεμένα αντικείμενα που θα συνδέονται με το δίκτυο των 5, της 5ης και 6ης γενιάς, 5G και 6G, αλλά δεν μιλούμε μόνο για το διαδίκτυο των δεδομένων. Θα έχουμε έξυπνε πόλεις, έξυπνα νοσοκομεία, ψηφιακά εργοστάσια, συνδεδεμένα οχήματα. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τεράστιο όγκο δεδομένων και θα προτείνουμε κάποιες λύσεις Ε, και φυσικά αυτά θα πρέπει να τα κρατήσουμε στην Ευρώπη για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από την καινοτομία και την πρόοδο. Να σας δώσω κάποια στοιχεία για να ξέρουμε τι, γιατί μιλάμε για την ανάπτυξη αυτών των συνδεδεμένων αντικειμένων που κάθε ένα αντικείμενο δημιουργεί περαιτέρω δεδομένα. Το 2030 θα έχουμε 500 ε, δις συνδεδεμένα αντικείμενα Τώρα έχουμε 7 με 8. Θα έχουμε τεράστιο όγκο δηλαδή δεδομένων ε, ενώπιών μας. Και θα πρέπει αυτά να τα προωθούμε σε επιχειρήσει, να τα προσανατολίζουμε για τι επιχειρήσει, παρόλο που θα είμαστε μια ανοιχτή ήπειρο και θα πρέπει και άλλοι να μπορούν να συνεισφέρουν τι τεχνολογίε του. Αλλά θέλουμε, θέλουμε να υποφεληθούν και οι δικέ μα επιχειρήσει. Και δεν θέλω να έχουμε μια προστατευτική προσέγγιση. Απλώς θέλω με πεφωτισμένο τρόπο να αγγίψουμε στο πρόβλημα και χωρίς αφέλεια. Εγώ ασχολούμαι με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, τις ε, νεοφυής και τις μεγάλες και θέλω να τις προστατεύσω στις, στην νέα μεταμορφωμένη, μετασχηματισμένη αγορά και να τις επιτρέψω να εγκληματιστούν και να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες για να κατακτήσουν και νέες αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αρχικά τις πέντε μέρες τεχνικής νοημοσύνης και παράλληλα θα έπρεπε να φέρουμε και μια νέα διάσταση για να μιλήσουμε για τη μεγάλη εφαρμογή αυτών των δεδομένων που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό θα είναι το δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσής μας που θα υποβάλουμε σε αρχές Μαρτίου. Οπότε, φτάνουμε ήδη σε επίπεδο εφαρμογών, τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε θέλουμε αξιόπιστα ε, στοιχεία που θα είναι φορείς των αξιών μας, γιατί θα καταλήξουμε τελικά σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό θα πρέπει να ελέγξουμε όλους τους κρίκους της αξιακής αλυσίδας. Θα πρέπει λοιπόν για να ελέγξουμε τεχνητή νοημοσύνη να γνωρίζουμε όλη την αλυσίδα ακόμη και τη γνώση και, την, και τον έλεγχο των δεδομένων. Γι' αυτό εγκύπτουμε στο θέμα για να έχουμε μια τεχνητή νοημοσύνη αξιόπιστη, ηθική, διοντολογική, υπεύθυνη, που θα ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας. Και κυρίως με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Οπότε σε αυτά τα θέματα α, α, προηγούμενε τις προηγούμενες μέρες ε, και την Λευκή Βίβλο χωρίς να σας τα αναφέρω εξονυχιστικά, θέλουμε να επικεντρωθούμε στη φύση των δεδομένων που θα τροφοδοτήσουν έναν αλγόριθμο, να δούμε ποια είναι αυτά τα δεδομένα, πώς συγκεντρώθηκαν, πώς συνδυάστηκαν, ε, είναι συμβατά με τον κανονισμό μας, ε, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όταν μιλούμε για θέματα διαστημικά, ή και για θέματα της καθημερινότητας. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε ε, για όλα αυτά, γιατί φυσικά θα πρέπει να είναι δεοντολογική η νομοθεσία, να συνάδει με τις αξίες μας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλη αυτή την αξιακή αλυσίδα προηγουμένως. Αυτή την προσέγγιση θα ήθελα να σας προτείνω, ώστε να υποφεληθούμε όλοι. Και αν επικεντρωθούμε μόνο σε αρχές που μιλούν για τι τελικέ εφαρμογέ τη τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα οι μεγάλοι όμιλοι θα ανταποκριθούν αμέσω, θα ασθενιστούν ε, αυτού του κανόνε, αλλά ίσω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θα έχουν την ευκαιρία να τι χρησιμοποιήσουν και θα προσκρούσουν σε φραγμού. Vous indiquez, on le détaillera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 Ε, ε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ε, διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή η δύναμη, το δυναμικό καθώς επίσης και ο υπολογισμός ε, έχει γίνει με διαφορετικό τρόπο στα ε, δίκτυα αλλά και στις ε, κεραίες. Ξέρετε ότι θα έχουμε πλήθος αντενών πλέον κεραιών και η διασύνδεσή τους θα είναι τελείως διαφορετική και οπωσδήποτε και οι συχνότητες θα είναι εντελώς διαφορετικές έτσι ώστε σε μικρές αποστάσεις να έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη ε, ροή. Και μετά έχουμε ε, και την ε, διαφορετική 5G, η οποία θα είναι σε πολύ περισσότερα GHz, έτσι ώστε να μπορέσουμε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα να κάνουμε μετάδοση δεδομένων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε εργοστάσια, σε μηχανήματα τα οποία θέλουν ακριβώς πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα όσον αφορά την ε, ε, μετάδοση των ε, δεδομένων. Εδώ πρέπει να μπούμε σε πολύ καλή θέση στην αγορά. Πρέπει να είμαστε οι πρώτοι. Το Κοινοβούλιο ήδη τον προηγούμενο Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, απέτησε από την Κομισιόν να μελετήσει το θέμα αυτό. Και υπάρχουν και χώρες μέλη οι οποίες επίσης πίεσαν. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω αυτήν την κοινή εργασία του Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Κομισιόν που που ε, λειτουργήσε μετά από παρένεση και του Κοινοβουλίου και κρατών μελών, ε, προτείνοντας ε, μία, πώς να το πω, όχι αρχιτεκτονική ακριβώς, αλλά μια αξιολόγηση κινδύνων. Έγινε αυτή η αξιολόγηση, έγινε αυτή η δουλειά. Ήδη από τον Οκτώβριο έγινε η σχετική ανακοίνωση και μετά οργανώθηκε και μια λεγόμενη εργαλειοθήκη έτσι ώστε ε, να δουλέψουν ε, τα κράτη με την σειρά τους. Η δουλειά βεβαίως έγινε εδώ από τις χώρες και η Κομισιόν μονάχα συντόνισε. Πρόκειται πραγματικά για κάτι ε, πρωτόφαντο. Δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να υπάρξει διαφοροποίηση. Θέλουμε μόνο να καθοριστούν, να οριστούν κανόνες. Θέλουμε όλοι οι operators να εμπλακούν ε, σε αυτήν την διαδικασία. Να σας πω επίσης ότι... Ε, έχουμε ε, ε, ο, πολλές βιομηχανίες οι οποίες είναι πραγματικά στην αιχμή του δωρατος ε, της τεχνολογίας, δεν θα πω ονόματα, αλλά πάντως κατέχουν και τα θέματα της έρευνας και τα θέματα του 5G και του εξοπλισμού. Απ' την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι όσον αφορά την εργαλειοθήκη θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε κάθε χώρα, σε κάθε operator να προχωρήσει. Βιομηχανική πολιτική είναι ένα θέμα απολύτως θεμελιώδου σημασίας. Το συζητάμε πολύ, το συζητάμε πολύ και μεταξύ μας. Το 2050 γιατί αυτός, αυτός είναι ο χρονικός ορίζον ε, της Πράσινης ε, Συμφωνίας. Το 2050 καταλαβαίνετε ότι ε, αλλάζει η γενιά, η βιομηχανία μας θα έχει... Α, δεν έχω άλλο χρόνο να τα πω πιο γρήγορα, λέει ο κύριος Μπλετών, να πω για θέματα όμως που ε, αφορούν το φάκελό μου και είναι τις αρμοδιότητες μου και είναι πολύ σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε την βιομηχανική στρατηγική. Υπενθυμίζω ότι έχουμε δουλέψει πολύ ανατομέα, έχουμε δουλέψει πολύ στο θέμα της αλυσίδας αξιών. Ε, η βιομηχανική στρατηγική βασίζεται και πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη φιλοδοξία της ε, Πράσινης ε, Συμφωνίας. Ε, μιλάμε για μία ολόκληρη γενιά θέλουμε ε, καθαρές ε, ενέργειες ε, προσβάσιμες και προσιτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Θέλουμε ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να ανταποκρίνεται στην Πράσινη Συμφωνία, αλλά και στην ανάγκη από την άλλη πλευρά καθαρής ενέργειας προσιτής για όλους και για τις βιομηχανίες ε, η πρόσβαση ε, σε, στις πρώτες ε, ύλες, κυρίως δε σε κρίσιμες πρώτες ύλες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως πρωτο καινοτομία, στην οποία αναφέρθηκα και πιο πριν. Ε, θέλουμε να ξαναεξετάσουμε και να βάλουμε σε νέες βάσεις όλη την αξία της παραγωγής, της μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, αλλά και στις μεγάλες επιχειρήσεις, ε, συνδεδεμένη και με την ε, στρατηγική των δεδομένων, συνδεδεμένες βεβαίως και με την ψηφιοποίηση και με τις τοπικές, περιφερειακές και άλλες ικανότητες η πόροι τώρα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά ε, τη, τους πόρους και τις ικανότητες στα πλαίσια του μετασχηματισμού. Η προστασία και στα πλαίσια της ε, Πράσινης Συμφωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Επομένως πρέπει να έχουμε έναν ε, μηχανισμό ε, ανάλυσης του άνθρακα στους, στις, στα σύνορα που θα προστατέψουν τις επιχειρήσεις μας, τις βιομηχανίες μας από εισαγόμενα προϊόντα που θα έχουν παραχθεί με διαφορετικό τρόπο και χωρίς την απαραίτητη προστασία. Όλα αυτά αφορούν τη βιομηχανική στρατηγική. Να πω και δύο λόγια πριν ολοκληρώσω ε, για την άμυνα και το διάστημα. Ε, θα έχω, ελπίζω, το χρόνο να σας μιλήσω άλλη φορά ε, για το θέμα της άμυνας επί του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει ε, συγκεκριμένη βούληση για δημιουργία ταμείου γιατί πραγματικά θα πρέπει η άμυνα να είναι κοινό θέμα για όλους. Θα βοηθήσει και θέματα κυριαρχίας και άλλα. Όσον αφορά δε το διάστημα Ξέρετε, ε, και για την άμυνα και για, την, ε, για το διάστημα ε, έχω κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν στα πλαίσια του επομένου ΠΔΠ. Ε, η διακυβέρνηση του ε, Γαλιλαίου είναι κάτι που μας απασχολεί, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Η εξέλιξη του Κοπέρνικου, επίσης ε, άλλες πρωτοβουλίες όπως το ε, και το SSA για την ασφαλή διαμετακόμιση στοιχείων, κυρίως μεταξύ κυβερνητικών αρχών. Επίσης, κυβερνό ασφάλεια. Ναι, ε, μου είχατε δώσει 15 λεπτά, 3,5 ε, λεπτά παραπάνω μίλησα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έκανα έτσι μια συνολική παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την γενική έποψη που μας δώσατε, για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία. Θα έχετε βέβαια και την, θα έχουμε και τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για θέματα ε, ε, αυτής της πολύ φιλόδοξης ε, βιομηχανικής πολιτικής. Ξέρω ότι όλα τα θέματα αυτά σας παθιάζουν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε και ξεχωριστή συζήτηση όταν θα έρθει ο δόκιμος χρόνος και όταν θα έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. 27 είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν τον λόγο, εκτός των συντονιστών, για πρώτη φορά Νομίζω ότι δεν θα έχουν όλη τη δυνατότητα να μιλήσουν. Ας ξεκινήσουμε πάντως με τους συντονιστές. Σε τρία λεπτά ο κάθε συντονιστής και μετά 7 λεπτά θα έχει ο, ο, ο κύριος Επίτροπος ε, στη διάθεσή του έτσι ώστε να απαντήσει ε, στους, ε, ε συντονιστές. Ο κύριος Έλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γερμανός από τη φύση μου και πολύ ενθουσιώδης ε, και στην Επιτροπή μας ε, πιστεύω αποφασίσαμε πολύ σωστά όταν σας δεχτήκαμε ε, ως Κοινοβούλιο για τη θέση του Επιτρόπου και χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Τρία ζητήματα. αφενός ε, κάτι πρακτικό. Πολλά από τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε ήδη αποτελούν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Διότι οι επικειμένες επενδύσεις ε, για πολλά αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με τα προγράμματα κοινοτομίας των ορίζοντα και άλλα. Και είναι σημαντικό και οι τρεις θεσμοί να κατανοήσουν καλύτερα πώς ε, θα γίνεται η αλληλεπίδραση, διότι διαφορετικά θα μας σταματήσουν οι ίδιες διαδικασίες. Για παράδειγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη ε, δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόταση του ΕΛΚ στην ε, διαπραγμάτευση. Οι σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσεις δεν συζητούνται. Επίσης, μιλάτε για περικοπές του προπολογισμού, ε, όπως γίνεται με την κβεντική τεχνολογία. Δεν έχουμε πια την κβεντική τεχνολογία, γιατί την ανέβαλε η Επιτροπή. Είναι λοιπόν ύψης της σημασίας οι τρεις θεσμοί για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα αυτές τις φιλοδοξίες, να κάνουν κάποιο προγραμματισμό, γιατί πολλά πράγματα πια δεν αναπόκειται μόνο στην Επιτροπή, αναπόκειται σε εμά και στη συνεργασία μας με το Συμβούλιο, το οποίο έχει δείξει ιδιαίτερο συντηρητισμό ε, στην διοργανική του λειτουργία και σε όλες τις ε, διαδικασίες. Δεύτερον, οι κανόνες ανταγωνισμού Όλοι αναφερόμαστε στο ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση των κανόνων ανταγωνισμού. Αλλά αν πας να δεις ε, πρακτικά τι γίνεται ε, στη δοκιμή καταλληλότητας, τι, τι, τι κάναμε. Ξεκινήσαμε τα αεροδρόμια, όχι με πράγματα που σχετίζονται με την πολιτική. Διαδικαστικά προχωράμε σε ελέγχους καταλληλότητας διετής ε, κάτι που έχει καθοριστεί ήδη στην ατζέντα. Η ατζέντα δεν εστιάζεται καθόλου στην βιομηχανική πολιτική ούτε σε θέματα κρατικής ενίσχυσης και σχεδιάζουμε σε 2,5-3 χρόνια από τώρα τη μεταρρύθμιση των, ε, κρατικών, ε, των εργαλείων κρατικών ενισχύσεων. Είτε πρέπει να επιταχύνουμε ή αλλιώς δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε φιλοδοξίες. Η τρίτη μου ερώτηση αφορά τα τεχνικά ζητήματα και τις προτεραιότητες ε, τις δημοσιονομικές και τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτών. Τώρα μιλάμε για IPCI, για το υδρογόνο, αλλά πρακτικά δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε μια εταιρική σχέση για το υδρογόνο που είναι κάτι διαφορετικό που ήδη διαπραγματευόμαστε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Θα ήταν να αποκτήσουμε μια εικόνα πώς θεσμικά μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε ρεαλιστικά να μπορούμε να ξεκινήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα το 2021, διότι διαφορετικά ε, θα βρεθούμε παγιδευμένοι στο αργό θεσμικό πλαίσιο και ενώ πολλά πράγματα έχουν αποφασιστεί κάπως διαφορετικά στο παρελθόν. Ευχαριστούμε κύριε Έλερ, ζητώ συγγνώμη για το χρονόμετρο. Είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ. η γραμματεία με βοηθά, αλλά τώρα το κατάλαβα, οπότε θα είναι σαφές ε, πόσο μπορούν να μιλήσουν οι συνάδελφοι. Ο κύριος Νέκα. παρακαλώ, ευχαριστώ. Δώστε μου τον ίδιο χρόνο, παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Επίτροπε Μπρετών, ήθελα να σας ε, καλωσορίσω και ήθελα να σας πω κατά την ακρόαση Αναφέρατε πολλές δεσμεύσεις που ξαναβλέπουμε εδώ στην παρουσίασή σας. Ήθελα να επιμείνω σε κάποια θέματα. Ε, βιομηχανική στρατηγική. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει να αντιμετωπίσει ένα stress test πολύ σημαντικό, διότι αφενός πρέπει να τηρούμε τι υποχρεώσει μα στο πλαίσιο τη Πράσινη Συμφωνία και από την άλλη πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ε, ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία. Να αποφύγουμε να φεύγουν οι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε ε, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μα ανησυχεί όσου ε, δραστηριοποιούμαστε στο βιομηχανικό κλάδο και αφορά το μέλλον μα. Άκουσα να λέτε για μέτρα, για μηχανισμούς προσαρμογής που θα εισαχθούν του χρόνου. Μήπως είναι κάπως ε, μεγάλη καθυστέρηση, μήπως θα επηρεαστεί αρνητικά ο κλάδος. Εγώ προέρχομαι από μια πόλη ε, όπου παράγεται, υπάρχει μεγάλη ε, σιδηρουργία και χαλιβουργία. Έχουμε πολύ χάλιβα που έρχεται από την Ουκρανία, την Τουρκία, την Κίνα. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντικές ζημίες στην ευρωπαϊκή χαλιβουργία. Επίσης θεωρώ ότι όσοι εργάζονται στον τομέα αυτό απογοητεύονται για τις βάσεις δεδομένων. Είπατε πολύ σωστά όσον αφορά τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών που πρέπει να τα προστατεύουν ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συμφωνώ απόλυτο και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, διότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από την κλοπή δεδομένων αυτή η κλοπή γίνεται περισσότερο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση και λειτουργεί ει βάρο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε μέτρα αποτελεσματικά, ούτω ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα ε, που βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος. Αυτό πρέπει να υποθεί πολύ καθαρά. Μετά, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, εξηγήσατε πολύ καθαρά ε, τι ε, θα υπάρχει προς χρήση όλων, ε, προς καθημερινή χρήση και πράγματα πιο εκλεπτισμένα. Το επικίνδυνο θα ήταν να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κακή, διότι κάποιο οπλισμένο ντρόν θα μπορούσε να περάσει πάνω από τα κεφάλια μας. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση, τη σωστή διάκριση και να ενημερώσουμε όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, διότι ήδη σημειώνουμε καθυστέρηση σε σχέση με τις ανταγωνιστικές μας χώρες και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση θα είναι τεράστιες οι απώλειες. Η κυρία Τζαμπάλοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Καλώ όρισατε κύριε Επίτροπε. Ελπίζω να είναι πολλέ οι συναντήσει που θα κάνουμε την επόμενη πενταετία. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε με την Κροατική Προεδρία εδώ στην Επιτροπή μα και σαφή προτεραιότητα τη Προεδρία είναι η ψηφιοποίηση. Το σχετικό θεματολόγιο και η διασύνδεσή της με το στόχο του πρασινίσματος της βιομηχανία και της ενέργειας. Αναφέρατε και τα δύο στην ομιλία σας. Η Πράσινη Συμφωνία ουσιαστικά βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του Κοινοβουλίου μέχρι στιγμή. Ε, είναι η λέξη που έχει αναφερθεί περισσότερο από όλες τις άλλες από τότε που ξεκίνησε η θητεία μας. Ωστόσο, στην άλλη πλευρά ε, στον αντίποδο υπάρχει η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και φυσικά και τα ψηφιακά ζητήματα μπαίνουν στην εξίσωση. Εάν δεν έχουμε ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή βιομηχανία και τη Ευρωπαϊκή οικονομίας δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε το κλίμα. Πώ μπορούμε λοιπόν να τα συνδυάσουμε αυτά πώ θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο, διότι όπω είπατε και εσεί στην ακρόασή σα, έχετε δεσμευτεί για μια νέα στρατηγική αναπτυξιακή για την Ευρώπη. Πώ σκοπεύετε να τη διασφαλίζετε σε συνδυασμό με την Πράσινη Συμφωνία. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε και επιμείνατε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και αναφερθήκατε ότι πρέπει να υπάρχουν ευνοϊκοί κανόνε για όλε τι επιχειρήσει ανεξαρτήτω μεγέθου πώς θα εργαστείτε εσωτερικά ούτω ώστε να μην πεταχτούν έξω από την εξίσωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί μιλάει, μίλησατε εσεί για τις εσωτερικέ διαδικασίες που έχετε εσεί ως Επίτροπος, Ωστόσο, οι εξωτερικές δράσεις θα μπορούσαν επίσης να σας καθοδηγήσουν στις εργασίες σας. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα αξίζουν την προσοχή μας, αλλά η πραγματική αξία θα προκύψει από το πώ θα αλληλεπιδρούν όλες οι διαφορετικές πολιτικές μεταξύ τους πολύ συχνά παρατηρούμε ότι απουσιάζει η συνέργεια μεταξύ διαφορετικών πολιτικών προτάσεων και δράσεων. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μαζί, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει τέτοια συνέργεια μεταξύ διαφορών πολιτικών. Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι κάτι που αναφέρατε εσεί. Αναφέρατε τι ε, ε, νεοφυεί επιχειρήσει, τι startups. Πώ μπορούμε να τι βοηθήσουμε, Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχουμε από τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι τις υποστηρίζουμε. Όλοι τις υποστηρίζουμε. Το έχουμε δηλώσει ήδη. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ε, συγκεκριμένα αυτά για τις ε, startups ε, για να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τζαβόλογο. Εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος Μάικλ Μπλός. Δεν είναι εδώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Είναι απολύτως σαφές οι στόχοι του Παρισιού θα επιτευχθούν μόνο με μια στρατηγική στρατηγική ο μετασχηματισμού της βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε μια έξυπνη λοιπόν βιομηχανική στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παραγόντες που αναφέρατε σήμερα, την ανταγωνιστικότητα, την πρόσβαση στους πόρους, την ενέργεια, τα δεδομένα. Παράλληλα, πρέπει να καταλάβουμε ότι μια πράσινη ε, στρατηγική βιομηχανική θα πρέπει να ε, είναι δεκτή μόνο αν οδηγεί στην ουδετερότητα την αν ε, επιτύχουμε τους στόχους στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας μέχρι το 25 και μέχρι το 30 ε, και δεδομένης της κλιματικής έκτακτης ανάγκης που εξήγηλε το Κοινοβούλιο και να τηρήσουμε επίσης και τους στόχους του Παρισιού. Και σήμερα δεν κατάλαβα εγώ καλά τι ακριβώς βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής σας, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλά τα πεδία της εργασίας σας εξαιρετικά ε, συναρπαστικά και δύσκολα, αλλά εσείς πώς το βλέπετε. Τέλος, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων πώς θα αξιολογηθεί, πώς θα αποτιμηθεί και επίσης σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού θεωρούμε ότι θα τα καταφέρει μόνο αν κάνουμε κάτι και με τη βαριά βιομηχανία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη χαλιβουργία, με την απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές ε, των ενεργοβόρων βιομηχανιών ε, των ε, μετάλλων όπως αλουμινίου, ε, της χαρτοβιομηχανίας και ήθελα να μου πείτε ποιους κλάδους και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα βοηθήσετε Ποια ευρωπαϊκή στρατηγική θα χρειαστεί, θα χρειαστεί ευρωπαϊκή στρατηγική, μπορεί να γίνει καλύτερη από ότι οι εθνικές στρατηγικές, τι καλό μπορεί να κάνει η Ευρώπη εδώ. Και μια δεύτερη ερώτηση, πολύ σημαντική. Πώ θα πάρετε του ανθρώπου με το μέρο σα για μια τέτοια διαδικασία μετασχηματισμού, του ενδιαφερόμενου δηλαδή, των μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι εταιρείε, του καταναλωτέ, του ανθρώπου που ζουν ε, στι περιφέρειε και που επηρεάζονται από, τις, ε, από τους μετασχήματους αυτούς. Πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι με το μέρος σας, διότι μια ε, τέτοια διαδικασία μετασχηματισμού θα γίνει αν έχετε στο πλευρό σας του οικονόμου, τους, τον οικονομικό κλάδο, τον οικολογικό κλάδο και τον κοινωνικό κλάδο. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ συναρπαστικά όλα αυτά που έχετε μπροστά σας. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η πολιτική θα δρά γρήγορα και αποτελεσματικά στο μετασχηματισμό της κοινωνίας για να γίνουν ε, οι αλλαγές για μια κλιματικά ε, ουδέτερη κοινωνία και οικονομία. Ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν για να μπορέσετε να επιδράσετε πάνω στην αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ο κύριος Παύλο Μπόρκεκ, εκ της Ταυτότητας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Στο Παρίσι πριν από μερικές ε, μέρες ε, κάνατε κάποιες ε, ρεαλιστικές δηλώσεις σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής του Κάπορτ Mechanism. Ecco, la Commissione sta parlando da, eh, πολύ σωστά είναι όλα αυτά και μάλιστα ε, και ο Επιτροπός και η και η ε, υπογράμμισαν το σύστημα ε, αυτό και φαίνεται να οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, ε, παρά αυτό το θετικό προήμιο, έχουν προκύψει και κάποιοι προβληματισμοί από τα όσα είπε η πρόεδρος Φοντερ Λάγεν στο φόρουμ στο Νταβός. Η πρόεδρος, ας πούμε, είπε ότι, θα υπή... ότι ενδεχομένως θα εγκατελειφθεί ο μηχανισμός αυτός μετά από τις προσπάθειες που φαίνεται να ξεκινά ε, και να αναλαμβάνει η Κίνα ε, έτσι ώστε να μειώσει το διοξίδιο του ε, άνθρακα. Ενδεχομένως η πρόεδρος Φοντερ σε συνεργασία με την καγκελάριο Μέρκελ φαίνεται λέω να ε, κάνουν ένα βήμα πίσω όσον αφορά αυτόν τον συνοριακό φόρο άνθρακα ε, πριν ακόμα αρχίσει να εφαρμόζεται. Επίσης ε, η Κομισιόν είχε πει ότι τέλος του 20 ή εν πάση περιπτώσει ένα χρόνο μετά θα άρχισε να εφαρμόζεται. Εν πάση περιπτώσει όμως λέω ότι μια πρόταση που ακόμα δεν έχει δει το φως να φαίνεται ότι ε, την παίρνουμε πίσω έτσι ώστε να μην αγγίξουμε τις ευαισθησίες άλλων παγκοσμίων ε, πρωταγωνιστών. Πάντως, ε, κύριε Επίτροπε, υπάρχει πραγματικά βούληση να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτός και αν ναι, σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ του ECR συντονιστής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Τέμσκι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, ήταν χαρακτηριστικό που το μεγαλύτερο τμήμα της ομιλίας σας ε, το αφιερώσετε στα ψηφιακά θέματα, που είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικά. Βλέπετε σε αυτή τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, κάποια θέση για την παραδοσιακή μας βιομηχανία τι ευκαιρίες θα έχει και η παραδοσιακή βιομηχανία, τι δυνατότητες ανάπτυξης, περαιτέρω ανάπτυξης στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε φιλόδοξους στόχους και γνωρίζουμε ότι από τη μια έχουμε το, τη Νέα Πράσινη Συμφωνία, το Brexit, σημαντικά, σημαντικό ρόλο και τμήμα στην οικονομία μας, στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης έπαιζε το Ηνωμένο Βασίλειο που, αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μας περιμένει ρηξικέλεθος μετασχηματισμός λόγω της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Και είχαμε και τις πρόσφατες προτάσεις της Φιλανδικής Προεδρίας που πρότειναν περικοπές ταυτόχρονα στο κοινοτικό προϋπολογισμό και στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε φιλοδοξίες μεγάλες, ταυτόχρονα περικόπτουμε τα κονδύλια. Επίσης, θα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που προτείνεται περικοπή στο ίμιση. Οπότε και οι πολιτικές ε, φιλοδοξίες ε, που συνδέονται με αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί θα έχουμε και πολλές δύσκολες προκλήσεις και ταυτόχρονα θα πρέπει να διαφυλάξουμε την βιομηχανία μας και την παραδοσιακή και όχι μόνο την καινοτόμα και την ψηφιακή. Δεύτερη ερώτηση αφορά αυτό το toolbox που είπατε, την εργαλειοθήκη. Γιατί γνωρίζουμε ότι στα θέματα αυτά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για την ασφάλεια, για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές, να τις γεφυρώσουμε. Γιατί και η καγκελάριος Μέρκελ είναι υπέρ της συνεργασίας με την Κίνα, για παράδειγμα. Δεν έχουν όλοι όμως την ίδια άποψη. Ευχαριστώ. Και τελευταίος συντονιστή, τελευταία συντονίστρια μάλλον, εκ μέρους της Γκουέ. κυρία Μάρκες. Απουσιάζει ο κύριος Μποτέγκα, θα την αντικαταστήσει μήπως. Όχι, οπότε κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για 7 λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συντονιστών και μετά ετοιμαστείτε γιατί 29 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για την υπόλοιπη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συντονιστές για τις ερωτήσεις τους. Η ερωτήση του κύριου Έλλερ πρώτα. Σίγουρα πολλά έγιναν αλλά θα πρέπει να δρέψουμε τους καρπούς και στις σχέσεις που θα έχουμε θα αλληλοβοηθηθούμε Επιτροπή Κοινοβούλιο και Κράτη-Μέλη. Και συμφωνώ με την κατεύθυνση που δώσατε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και υπάρχουν και κάποια προγράμματα που δεν υπάρχουν στο ΠΔΕΛΤΑΠΗ και που μας προβληματίζουν. Το Ταμείο Άμυνας, για παράδειγμα. Το Μανιφέστο για την κβαντική υπολογιστική. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και να επαγρυπνούμε στη διαπραγματεύση ώστε να λειτουργήσουμε τα υπάρχοντα και να έχουμε προϋπολογισμό που θα σταθεί στο ύψος των φιλοδοξιών μας. Και σε ό,τι φορά την ανταγωνιστικότητα Ευχαριστώ που το επιθυμήσατε γιατί είναι κέρια σημασία και στην επιστολή ανάθεση καθηκόντων και τη δική μου και τη κυρία Φεστέγκερ. Αυτό ακριβώ λέμε ότι θα πρέπει να προταθεί. Και εγώ ασχολούμαι με το θέμα αυτό και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στους κανόνες του ανταγωνισμού και πώς θα ενταχθούν αυτά νέα βιομηχανική στρατηγική. Και αυτό αποτελεί επιθυμία και των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου πιστεύω και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξουμε, να εξελιχθούν αυτοί οι κανόνες ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη και τη Νέα Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση αλλά και το γεωπολιτικό χαρακτήρα της Επιτροπής ε, στα πλαίσια των νέων, του νέου σχετισμού δυνάμεων που δημιουργείται. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, IPCI. Σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα όπως το υδρογόνο για τα οποία θα πρέπει να έχουμε κάποια σχέδια να τα αναπτύξουμε. Έχω και άλλες ιδέες. Σημαντικό αυτό το εργαλείο των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει και εκεί να σπεύσουμε όμως. Και μάλιστα στα πλαίσια της βιομηχανικής μας στρατηγικής θα συζητήσουμε από κοινού τα πιο μακρόπνοα, πιο μεγάλη επιβολα σχέδια για τα οποία κρίνουμε απαραίτητο τον συντονισμό μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, κρατών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως προς αυτά συμφωνώ επίσης μαζί σας. Ο κύριος Νίκα ήταν ο δεύτερος συντονιστής που μίλησε. Για τη βιομηχανική στρατηγική, φυσικά σημαντική είναι η ανταγωνιστικότητα, ο ανταγωνισμός. Θα πρέπει να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε τις μετεγκαταστάσεις να μην χάνουμε τη βιομηχανία μας και ο συνοριακός φόρος του άνθρακα είναι τμήμα της Νέας Πράσινης Συμφωνίας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση να τον μειώσουμε ή να τον καταργήσουμε. Η φιλοδοξία είναι δεδηλωμένη και η πρόθεση και μάλιστα έτυχε και τη υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα εφαρμοστεί αυτό ο συνοριακός φόρο άνθρακα, ο μηχανισμό προσαρμογή του άνθρακα στα σύνορα. Και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Και εγώ θα προωθήσω την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Για κάποιου τομεί, τη χαλιβουργία, τη τσιμετοβιομηχανία, θα είναι από τα πρώτα θέματα, του πρώτου τομεί που θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, ώστε να λάβουμε άμεση δράση. Μιλήσατε και εσείς για τα δεδομένα. Είπατε ότι θα ήταν προτιμότερο τα, τα περισσότερα, αν όχι το σύνολό τους, να αποθηκεύονται και να τη επεξεργασία στην Ευρώπη. Και αυτό το θέμα θα το αναφέρουμε στην στρατηγική μας για τα δεδομένα. Μαρτίνα Τζαμπαλόβα μιλήσατε για τη Νέα Πράσινη Συμφωνία και την ανάπτυξη. Η ελληνική καμπίνα κατέρευσε. Ε, θέλουμε μία ισορροπημένη στρατηγική, μία στρατηγική άμυνα ταυτόχρονα. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια σημεία και είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας που ενδιαφέρει τους πολίτες ε, και να αυξήσουμε και την παραγωγικότητα γιατί αν θέλουμε η ανάπτυξή μας ε, να προχωρήσει κάτι που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και σε, έναν, ε, σε μια ήπειρο με σχετικά σταθερό πληθυσμό θα χρειαστεί αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό ενδιαφέρει και είναι τίμα της βιομηχανικής μας πολιτικής. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Και έχουμε εδώ ένα χρονικό ορίζοντα 25 ετίας. Δεν θα πρέπει να γίνει ε, εν μία, δεν θα μπορεί να γίνει εν μία νυχτή. Και ορίσαμε τα 25 χρόνια αλλά θα πρέπει από τώρα να ανασκουμποθούμε και να στρωθούμε στη δουλειά, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα αναπτύξουμε κάποια εργαλεία, κάποιες νέες τεχνολογίες, κάποιες νέους τρόπους παραγωγής και θα αυξήσουμε έτσι και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά μας. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κέριο ζήτημα και βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής μας και του μυαλού μου. Θα πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη θέση στην αξιακή αλυσίδα και για όλη την βιομηχανική στρατηγική και για την κυκλική οικονομία. Είναι σημαντικό τα προϊόντα που θα αναπτύξουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο στόχο και θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη ε, αντιμετώπιση αυτού του θέματος, προϊόντων και υπηρεσιών. Και επίσης όλα αυτά που αφορούν τη σχέση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ομίλων. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Αυτά και άλλα πολύ σημαντικά θέματα θα ενταχθούν στη στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τελευταίο θέμα το οποίο αναφερθήκατε είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup. Βεβαίως η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικά μια ενιαία αγορά, μια ενοποιημένη αγορά ε, εγώ θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, ε, να δω ακριβώς ποιες είναι, ε, ποια θα είναι η καλύτερη πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Βασιστείτε πάνω μου, πραγματικά εγώ θέλω να αρθούν όλα τα εμπόδια και οι φραγμοί που δυσκολεύουν την εξέλιξη των νεοφιών επιχειρήσεων και τα θέματα τα οποία αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία βεβαίως θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό όσον αφορά ε, την ε, κυρία που μίλησε εξ ονόματος των Πρασίνων. Πρέπει να πω ότι και στο θέμα που θίξατε η στρατηγική είναι σαφής. Είπατε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή στρατηγική και με ρωτάτε ε, γιατί είναι καλύτερα να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Μα κοιτάξτε, όσο ε, ε, πρόκειται για στρατηγικές οι οποίες ξεπερνούν τα σύνορα, επομένως χρειαζόμαστε φιλοδοξία η οποία να είναι σαφώς ευρωπαϊκή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε την υποστηρίζει το σύνολο των κρατών μελών. θα εμπλακούν ε, τα, ε, ε, οι άνθρωποι. Ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει ανθρώπινη διάσταση σε αυτό που λέτε. Όμως τώρα υπάρχουν και πολλές περιφέρειες οι οποίες θα είναι παρούσες όσον αφορά την δίκαιη μετάβαση και θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Επίσης, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι μιλάμε για 25 χρόνια διάρκειας, άρα μιλάμε για μία γενιά, άρα θα πρέπει να ε, βρούμε, να σκεφτούμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, τα οποία θα δώσουν τα καλύτερα ε, αποτελέσματα, ενδεχομένως ομόλογα, μεγάλης διάρκειας ορίμανσης και μηδενικό ενδεχομένως επιτόκιο. εάν μέσω του μηχανισμού ε, μπορούμε να έχουμε και του, του, του μηχανισμού ε, προσαρμογής ε, στα σύνορα, αν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα καλό εργαλείο, μπορούμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, όσον αφορά αυτό το συνοριακό φόρο άνθρακα, δεν ε, ε, υπάρχει περίπτωση οπισθοχώρησης όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, πρόκειται για απόφαση η οποία υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο και φυσικά και από το Κοινοβούλιο και εδώ δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε μέτρα για να υποστούν κάποιοι άλλοι διακριτική μεταχείριση, αλλά ε, είναι, θέλουμε ε, όλοι να ξεκινούν από ένα ίδιο επίπεδο. Θέλουμε όλοι να εφαρμόσουν αυτήν την ε, πρακτική, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα όπως θα Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις βιομηχανίες μας. Κύριε Δεν ε, αναφέρθηκα στις μη ψηφιακέ ε, βιομηχανίες. Ε, θα ήθελα, αλλά δεν είχα χρόνο. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είχα προβλέψει να αναφέρω. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι βιομηχανίες αυτές αντιπροσωπεύουν το 24% της δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς δεν θέλουμε, δεν έχουμε δηλαδή την άποψη ότι ε, το ψηφιακό θα κατακλείσει τα πάντα και θα αντικαταστήσει τα πάντα. Υπάρχουν ε, ε, άλλα στοιχεία όπως είναι η παραδοσιακή διάταξη, όπως είναι οι σχέσεις με τους καταναλωτές, με τους πολίτες. Αυτά όντως θα εξελιχθούν, θα κινηθούν, θα μετακινηθούν. Αλλά παρόλα αυτά δεν μιλάμε μόνο για ψηφιακά. Όσον αφορά τα, το αμυντικό σύστημα, ε, εδώ έχουμε το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ε, και εγώ θα ήθελα να συμμετάσχουν όλες οι χώρες ε, και τολμώ να ελπίσω ότι σιγά σιγά και με τα χρόνια που θα έχουμε προοδεύσει θα έχουμε και κάποια στρατηγικά προγράμματα πάντα στα, με γνώμονα την κυριαρχία μας και θέλουμε όλοι να συμμετάσχουν και τα λέω όλοι, αναφέρομαι στις επιχειρήσεις ε, ανάλογα με το μέγεθός τους αλλά και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δηλαδή δεν θα είναι μόνο για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Και βεβαίως πιστεύω ότι όλοι θα έχουμε ενδιαφέρον και συμφέρον να επιλέξουμε την ευρωπαϊκή οδό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ήμουν όσο αυστηρό θα ήθελα. Μιλήσατε περισσότερο, ωστόσο είναι πολλέ ενδιαφέρουσε ε, ερωτήσει τι οποίε πρέπει να απαντήσετε. Δεύτερο γύρο, ίσω θα, ε, θα μα δώσουν και οι διερμηνεί 15 ε, λεπτά επιπλέον. Αλλά παρόλα αυτά να μην ξεπερνάτε το ένα λεπτό ο καθένα, έτσι ώστε να μπορέσει και ο Επίτροπο να απαντήσει και ίσως να κάνει μια γενική απάντηση, όχι να απαντήσει σε καθένα χωριστά. Αυτό είναι αδύνατο. Ο πρόεδρος Μπούζεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτρόπη που βρίσκεστε εδώ. Our industrial independence. Αναφέρνετε ε, βιομηχανική στρατηγική και βιομηχανική αυτονομία. Έχουμε τη χαλιβουργία η οποία από τη ΚΟΚ. Και καμία τεχνολογία δεν μπορεί να το αντικαταστήσει σήμερα αυτό. Και από αυτό εξαρτώμαθα ω Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία. Έχουμε τεράστια χαλιβουργία και είναι αναγκαίο να εισαχθεί κάρβουνο από τη Μοζαμβίκη, από την Κίνα, από τη Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να διατηρηθεί αυτό το υλικό, το κοκ, στη λίστα των βασικών πρώτων υλών. Και αυτό εξαρτάται από τη δική σας απόφαση, ε, κύριε Επίτροπε. Οπότε ε, ελπίζουμε ότι θα διατηρήσετε το κάρβουνο και το ε, κοκ στην, στον κατάλογο. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόια, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα μιλήσω Ιταλικά. Δύο θέματα Πρώτον, μεταξύ πράσινη συμφωνία και βιομηχανία, κάποιοι λένε θα την πληρώσει η βιομηχανία, αλλά λένε θα είναι ευκαιρία. Εγώ πιστεύω ότι είναι αναγκαίο, διότι εγώ, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι εμεί δεν θα επιτύχουμε του στόχου ε, τη απαλλαγή από τι ανθρακούχε εκπομπέ, αν δεν κάνουμε ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα όσον αφορά ε, τις πρώτες ύλες, ε, τις ενεργειακές, ε, την προσαρμογή των επιχειρήσεων μας, των, μεταφορών κτλ. Πώς θα κάνουμε αυτό το τεχνολογικό άλμα που απαιτείται για τους στόχους αυτούς ε, μέσω της έρευνας, της καινοτομίας ε, στις επιχειρήσεις αλλά και μέσω μιας βιομηχανικής πολιτικής που θα πρέπει να συνδυάζει με τη συνέργεια όλα αυτά τα στοιχεία και φυσικά να μην εμποδίζουμε και την ενίσχυση ορισμένων φορέων ε, που επεξεργάζονται δεδομένα σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους διότι η στρατηγική αυτή που αποδυνάμωσε τους καλύτερους από εμάς δεν θα μας δώσει καλά αποτελέσματα και δεν θα συμβάλλει στην απαλλαγή από ανθρακούς εκπομπές. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκρούλερ από το Ρινιού. Κύριε Επίτροπε, ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τις δηλώσεις σας όσον αφορά τις πολιτικές σας προτεραιότητες. Μιλάτε πολύ καθαρά Είστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας ισχύρης και ανταγωνιστικής. Ε, λέτε στους Αμερικανούς και τους Κινέζους ότι για να κάνουν δουλειά στην Ευρώπη πρέπει να ε, τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, και όπως είπατε έχει έρθει η ώρα να σταματήσει η Ευρώπη να είναι αφελής. Συμφωνώ μαζί σας, ο ψηφιακός κλάδος, τα δεδομένα μας, οι συνδέσεις μας, οι οπτικές σύνες, οι δορυφορικές συνδέσεις και η κυβερνοπροστασία είναι πλέον ένα απόσπαστο κομμάτι και βασική κλάδη για την στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν τον ελεγχό του. Στι 4 Μαρτίου θα παρουσιάσει τι μεγάλε γραμμέ τη μελλοντική βιομηχανική στρατηγική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί τι θεωρείτε για ένα, μια ευρωπαϊκή πράξη για του ε, ε τομεί που συμμετέχουν ε, στην αυτονομία τη Ευρώπη, στο διάστημα, στην ασφάλεια, ε, στην αεροναυτική. Στην αεροναυτική. Ευχαριστούμε, κυρία Καρβάλιο, ε, συντονίστρια του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, μερικοί κλάδοι όπως η βιομηχανία, η βαριά βιομηχανία, είναι πιο δύσκολο να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές, ε, σημαντικοί κλάδοι για τη βιομηχανία. Ενεργοβόρες βιομηχανίες, χαλιβουργία, ε, η επεξεργασία προϊόντων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πραγματική επανάσταση τεχνολογική. Θέλουμε έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, δημιουργία προτύπων. Πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο κατωμερών, αλλά και για να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσει αυτά. Ο κύριο Ροπ, Ροπέ, συγγνώμη, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο φιλόδοξο έργο σας και κατάλαβα από την ε, αρχική σας ομιλία ότι πιστεύετε πως για τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να είμαστε το ίδιο απαιτητικοί με τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη και παράγονται εδώ. Και αυτό δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν, αλλά και την διαδικασία παραγωγής, τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα πρέπει και για τα εισαγόμενα προϊόντα να ισχύουν οι ίδιες αυστηρές προδιαγραφέ και πρότυπα που ισχύουν για τα δικά μας προϊόντα, τα ενδοευρωπαϊκά. Θα πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη τι κλιματικέ αλλαγέ. Όταν σκεφτόμαστε τι, παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγαθών σε τρίτε χώρε, σίγουρα κάτι τέτοιο δεν συνάδει με του κλιματικού μα στόχου. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στι εισαγωγέ. Πρόκειται να υποβάλλετε σχετικέ προτάσει. Ευχαριστώ, κύριε Άλβαρες Μονιό. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι τις πρώτες 100 μέρες εσείς και η κυρία η Επίτροπο Σπεστάκη θα υποβάλλεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχετε σκοπό να εμπλέξετε σε αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριο Έλερ σα μίλησε για τη βελτίωση επικοινωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πώ σκοπεύετε συγκεκριμένα να αναμίξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα από την αρχή, από τι πρώτε 100 μέρε Επίση, ε, θα συμπεριλάβετε και τη διάσταση του φίλου σε όλα αυτά. Γιατί στο σχέδιο της Λευκής Βίβλου ε, που άρχισε να κυκλοφορεί δεν είδα τίποτα για το φίλο και τη συνεκτίμηση της διάθεσης του φίλου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριανό από την ταυτότητα και δημοκρατία. Όχι. Μπάρενσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω Ολλανδικά γιατί θα χρησιμοποιήσω δύο Ολλανδικά παραδείγματα. Μία εταιρεία μας ε, ζήτησε εξαγωγική άδεια για εξαγωγή τεχνολογικών ε, τμήματων και η Κίνα ασκεί πιέσει ε, στην Ολλανδική κυβέρνηση, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε ασκούν ε, αντίρροπες πιέσεις σε σχέση με τις Κινέζικες. Πώς ε, θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτή την, την διαμάχη Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω ούτε από την ΕΠΑ ούτε από την Κίνα και έχουμε πολλές αφιβολίες για τις κρατικές ενισχύσεις που δίνει η Κίνα στη βιομηχανία της. Πώς θα διαμορφώσουμε τη βιομηχανική μας στρατηγική ώστε να προστατέψουμε την βιομηχανία μας ιδιαίτερα από τον αθέμητο ανταγωνισμό τρίτων χωρών γιατί αν θέλουμε μια ειφορία στη βιομηχανική μας πολιτική και διαφύλαξη της βιομηχανία μας θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σρό από το ECR. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρετό, μιλήσατε για την 5G γενιά, την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα. Μιλήσατε για ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει όμως για να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία μας να είναι και προσιτές οι τιμές της ενέργειας. Ε, να λάβουμε υπόψη και εναλλακτικέ πηγές όπως το βιοκαύσιμο. Πριν από μία εβδομάδα στον Ταβός αναφέρθηκε ότι θα καταργηθούν κάποιοι κανόνες προκειμένου να προωθηθούν συγκεκριμένες μορφές ενέργειας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις υποσχέσεις της ε, Επιτρόπου Φόντερ Λάιεν. Θέλετε η βιομηχανία μας να είναι και κερδοφόρα και όχι μόνο φιλοπεριβαλλοντική. Ο κύριος Ζωρίνιο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κυρία Φοντερ Λάιν χαρακτήρισε γεωπολιτική την Επιτροπή. Γι' αυτό όμω χρειάζεται και τα απαραίτητα εργαλεία και του μηχανισμού για να είμαστε ένα αξιόπιστο ε, παράγοντα ε, στο διεθνέ προσκήνιο υπέρ μια ε, ανθρωπιστικής ανθρωπιστική και βιώσιμη παγκοσμιοποίηση. Έχουμε το πρόγραμμα και τη διαστημική μας, για τη διαστημική μας πολιτική, για το οποίο όμω και ο και για τα δύο προγράμματα που παρακολούθησε είχαμε μια υπερκομματική ε, έκτακτη πραγματικά άνευ προηγουμένως συνεννόηση, αλλά δεν έχουμε αρκετά κονδύλια. Και για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, η Φιλανδική Προεδρία πρώτη ε, περικοπές, διέλυσε ουσιαστικά το πρόγραμμα ε, Ψηφιακή Ευρώπη και για την διαστημική πολιτική επίσης πρότεινε κάποιες περικοπές. Πώς ε, θα μπορέσετε εσείς να συνδυάσετε τα δύο προγράμματα ώστε να μην ε, υποστούν σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πεκάρινεν. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Στην ε, Ευρώπη η βιομηχανία μας εξαρτάται ε, από πρώτες ύλε που εισάγονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα σπάνια μέταλλα, ας πούμε, είμαστε εξαρτημένοι κατά 90% από την Κίνα. Θέλουμε να προωθήσουμε, ας πούμε, τα ηλεκτρικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, αλλά εμείς παράγουμε πολύ λίγα από ε, τα, ε, ε, τις ύλες που χρειάζονται όπως το κοβάλτιο ή οποιαδήποτε ε, άλλη. Επομένως, η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτό είναι αλλη επομενως η ερωτηση μου ειναι η εξης αυτο ειναι κατι που σας φοβίζει, αποτελεί μία από τις προτεραιότητές σας. Ευχαριστώ κυρία Βάης, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ούρσουλα Βαντελάιεν τον Ιούλιο είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την αχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας. Διαβάζοντας ε, τα νέα του ε, Digital Europe, ε, αναφέρονται δύο προβλήματα όσον αφορά το ε, ψηφιακό προφίλ της Ευρώπης που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουμε και για το εμπόριο και για τις μικρομεσαίες και ε, για το κλίμα. Λείπουν 900.000 θέσεις εργασίας ε, για, ε, που πρέπει να πληρωθούν από άτομα με ψηφιακές ικανότητες. Τι θα κάνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας για να καλύψω το κενό αυτό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρει η Digital Europe. Σχεδόν το μισό από τις θέσεις εργασίας γενικώ χρειάζεται περισσότερες ε, ε, ικανότητες χρήσης ενός ψηφιακού, μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης που θα δώσει περισσότερες δυνατότητες κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mr. Commissioner, thank you. I want to ask a question. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, σχετικά με την ε, στρατηγική δεδομένων. Είπατε ότι θέλετε ε, να γίνει προτεραιότητα η αποθήκευση των δεδομένων στην Ευρώπη. Πώς θα το κάνετε αυτό. Ε, γιατί οι περισσότερες υπηρεσίες έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ε, υπογραμμίζεται την ανάγκη ε, ανταλλαγής μη προσωπικών ανωνύμων δεδομένων στην βιομηχανία. Αυτό όμως μας οδηγεί σε κάποιο δίλημα τι γίνεται όταν ε, υπάρχουν ε, κάποιοι operators οι οποίοι διακρατούν πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων στοιχείων. Ε, πώς θα ξεπεράσετε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σολισπέρες, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, ερευνητέ, έχουμε επιχειρηματίε, έχουμε ικανότητε. Ωστόσο, οι νέε επιχειρήσει και οι νεοφυεί αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ε, ανάπτυξη και γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά και γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Ε, ε, επίσης, πολλές ε, εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ψάχνουν άλλα οικοσυστήματα καινοτόμα που όπου θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να εξελιχθούν. Ε, πηγαίνουν πολύ συχνά προς τις ΗΠΑ όπου το κεφάλαιο κινδύνου αντιμετωπίζει τελείω διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε όμω ανθρώπινο κεφάλαιο και κεφάλαιο καινοτομία. Τι θα κάνετε στα πλαίσια αυτή τη βιομηχανική ε, στρατηγική και τη στρατηγική για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι θα κάνετε έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα που έχουν ε, οι μικρέ επιχειρήσει και οι startups έτσι ώστε να γίνουν scale-up. Τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτές οι εταιρείες να μείνουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΕΛΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός ε, Τιμπίλιους. Έχετε δίκιο κύριε Επιτροπέ, τα δεδομένα είναι το μέλλον μας. Και πρέπει να χρησιμοποιηθούμε σωστό τρόπο. Δύο ερωτήσεις έχω. Εκτός των ε, δεδομένων υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αναπτύσσονται ας όπως η επεξεργασία του γονιδιώματος ας πούμε ε, και επίσης η εξέβρεση νέων εργαλείων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όμως ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται ένα σωρό πράγματα τα οποία επιτρέπονται ήδη σε μέρους πολιτής και στην Κίνα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό για την Κεντρική Ευρώπη, για τις χώρες της Βαλτικής. υπάρχουν ας πούμε ζητήματα τα οποία αποφασίζουν στην Ευρώπη όπως το Global Europe. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα ε, κάποια εξειδικευμένα ας πούμε προβλήματα ε, ή ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα επιβραδύνουν την ε, εμπλοκή μας. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιφερειακά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τότου. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή Ήτρε. Κατά την άποψή μου, η ρομποτική και άλλες ε, ε, υπηρεσίες που, που έχουν στόχο τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων ε, προϊόντων είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία και για την κοινωνία. Πιστεύω ότι τα καλά παραδείγματα είναι ας πούμε τα παραδείγματα των έξυπνων σπιτιών. Θα πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες που αυτές οι νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα δίνουν και η ανάπτυξη τεχνολογιών κατά την ε, κατεύθυνση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Κομισιόν ε, με χρηματοδότηση και στοχευμένα προγράμματα να δώσει τη δυνατότητα χρήσης αυτών των τεχνολογιών από όλους τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις. Κατά την άποψή σας ή μάλλον ποιες επιπλέον δράσεις προτίθεται η μαλλον ποιε επιπλεον δρασεις Επιτροπή να λάβει έτσι ώστε να αναπτύξει, να μεγαλώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κουταζάρα, πρόεδρε, και καλώ ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που αναφέρατε τα σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη και την αξιοπιστία τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντική η τεχνολογία. Θα μα βοηθήσει ε, επίση να αντιμετωπίσουμε και τι προκλήσει που θα προκαλέσει. Και εδώ αναφέρομαι στι ανισότητε που θα προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη, τα στερεότυπα του φύλου και τις ανισότητες στην αγορά επίσης. Οπότε θέλω να μου πείτε τι σχέδια έχετε για να αντιμετωπίσετε όλα αυτά επίσης. Θα ήθελα να αναφερθείτε στο χρήση των δεδομένων ως δημοσιογαθού. Και ήθελα να σας ρωτήσω επ' αυτού, με ποιο τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε επικοδομητική συνεργασία στον τομέα των δεδομένων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φόρων, ώστε να αποφύγουμε το σύστημα δεδομένων ε, να οδηγήσει σε ανισότητε και σε κατάχρηση των δεδομένων και σε υπερβολική συγκέντρωση δεδομένων σε συγκεκριμένα μέρη. Ευχαριστούμε ο συνάδελφο κύριο Άντρεσεν. Ευχαριστώ κύριε Μπρετόν. Είμαι εισηγητή ε, για το Κέντρο Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και ήθελα να σα ρωτήσω για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα η κυβερνοασφάλεια για τα επόμενα χρόνια. Όπω έχουν όμως τα πράγματα σήμερα, οι απαντήσεις που λαμβάνουμε δεν είναι ικανοποιητικέ. Θα ήθελα να μου πείτε τι σχέδια έχετε για την κυβερνοασφάλεια γενικότερα. Κάποιε ιδέε ε, και νομοθετικές έχετε για την κυβερνοασφάλεια και σε σχέση με το κέντρο κυβερνοασφάλειας ήθελα να μου πείτε τι σχέδια έχετε για το κέντρο. Ξέρετε υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία μεταξύ κάποιων κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια λύση ώστε να προχωρήσει το κέντρο κυβερνό ασφάλεια. Θέλω να μου πείτε τι σχέδια έχετε γι' αυτό. Thank you very much, Eva. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καηλή. Thank you. Um, so... Ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος μας μεταμορφώνεται και αλλάζει. Και ήθελα να μου πείτε, κύριε Επίτροπε, μετά από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχουμε ε, στο επίκεντρο τα δεδομένα, ε, και η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει και σε προστατευτισμό. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον προστατευτισμό. Ε, παρατηρούμε έναν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Κάποιες ε, χώρες χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να υποστηρίξουν αυτόν τον προστατευτισμό. Θέλουμε παγκόσμια δεδομένα τώρα για τη χρήση των δεδομένων, όπω κάνουμε και για τη κίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων. Πώ θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το παράδοξο. Και επειδή χρειαζόμαστε και όραμα και ηγεσία για να είμαστε σημαντικοί παγκοσμίω και ανταγωνιστικοί, πώ μπορούμε να το επιτύχουμε, να εξισορροπήσουμε δηλαδή ε, τις αγορές με τους ανθρώπους, ε, την προστασία του απορρίτου που είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας μας ε, και ταυτόχρονα εξορισμού να έχουμε ε, υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα καταπνίξουν την καινοτομία. Δεν είναι εύκολο. Και χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ, γιατί έχετε τις γνώσεις και είμαι βέβαια ότι θα βρούμε λύσεις. So much. Ε, Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Σαλένη. Ευχαριστώ. Τρία σημεία. Πρώτον, όσον αφορά το συνοριακό φοροάνθρακα. άνθρακα, ο carbon tax, ε, είναι ένα μέτρο απαραίτητο υπό μία προϋπόθεση ότι δεν θα είναι η εναλλακτική προς το ETS αλλά ότι θα συνεπάρχει διότι αλλιώς τα θετικά αποτελέσματα για τη βιομηχανία μας θα ακυρωθούν τελείως θα πάψουν να υπάρχουν τελείως το δεύτερο πολύ σημαντικό εσείς ε, πιστεύω έχετε ένα πολύ βασικό καθήκον το να αντισταθμίσετε να εξισορροπήσετε μάλλον τη νομική προσέγγιση της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για το αντιτράστα. Εμείς ε, έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να προστατευτούν και ένα από τα εργαλεία για την προστασία τους είναι να μην καταστρέψουμε τη μεγάλη μας βιομηχανία. Τρίτο σημείο για το διάστημα. Για το διάστημα εσείς πρόσφατα υπενθυμίσατε ότι είναι αναγκαίο να αλλάξει η διακυβέρνηση και συμφωνώ μαζί σας. Ωστόσο, έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει για την διακυβέρνηση. Σε ποια σημεία μπορούμε να παραμείνουμε μαζί και δεν αναφέρομαι τώρα στον προπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση στα γαλλικά. Κύριε Επίτροπε, έχετε αναλάβει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο για τη βιομηχανία, το διάστημα, την άμυνα. Είναι τεράστιο αυτό το χορτοφυλάκιο και παρουσιάζει και προβλήματα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόβλημα χρηματοδότησης, το πρόβλημα του Brexit, διότι η Μεγάλη Βρετανία βγαίνει από την Ένωση. Ήταν σημαντική στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η ερώτησή μου είναι πώς θα... τι θα κάνετε για την αντίσταση που δείχνουν κάποια κράτη-μέλη που συχνά αναφέρεται στα άρθρα 3, 4 και 6 της ε, το 346 ε, της συνθήκης ε, που αναφέρεται στον τομέα της προστασίας και της άμυνας και της ασφάλειας και τα μέτρα που παίρνουν τα κράτη-μέλη. Τι θα κάνετε λοιπόν για να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντική στην Ευρώπη, δηλαδή και η αγορά αμυντικού εξοπλισμού με διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς πραγματικούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα πέντε συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους. Κύριε Κούπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να αναζωογονήσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Και να μην αυτό ο εξορροπητικός παράγοντας της βιομηχανίας. Επίσης θέλουμε ψηφιακή οικονομία, δεδομένα. Μιλάμε πολύ για το 5G, αλλά θέλουμε και νέες ε, υποδομές. Πώς θα ανοίξουμε την όρεξη των χρηστών, λοιπόν, ή και των, ε, των ε, εταιριών τηλεπικοινωνιών να επενδύσουν ταχύτερα. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μείνει πίσω και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για το φάσμα το 5G. Μερικές χώρες δεν έχουν καν αρχίσει, ενώ άλλες έχουν ξεκινήσει τις δοκιμές. Επίσης, η οικονομία των δεδομένων ε, θα πρέπει να συνδυαστεί με την καινοτομία, τις καλύτερες ενεργειακές λύσεις, το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Θα τα καταφέρουμε όμως χωρίς υποδομές. Αυτόματα θα αφήσουμε τις άλλες υπήρους να ηγηθούν, αν δεν το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και υπάρχει και το θέμα το οικονομικό. Είναι κρίμα 6,6 δις να τα δίνουμε στους δορυφόρους και να αγνώμα το θέμα του φάσματος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν σας ευχαριστώ που ήρθατε. μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις δοκιμές, του τεστ για την τεχνητή και τα data sets ε, για να αποφύγουμε τις διακρίσεις. Πώς θα, θα ενεργήσετε. Επίσης, τα κράτη-μέλη δημιουργούν μεγάλη ποσότητα δεδομένων, αλλά δεν υπάρχει κάποια συστηματική προσπάθεια για τη δημοσίευση αυτών των δεδομένων, ώστε να είναι αναγνώσιμα από μηχανές. Πώς θα εναρμονίσουμε την παραγωγή των δεδομένων, ώστε να γίνει καλύτερη και πιο εύχριστη η χρήση τους στις δοκιμές για τη τεχνητή νοημοσύνη. Κυρία Μάρκες, έχω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομες κύριε Επίτροπε. Η πρώτη αφορά τους κοινούς χώρους δεδομένων. Πώς θα τους οργανώσουμε. Για ποιο τομέα θα είναι ο πρώτος τέτοιος κοινός χώρος. Η υγεία έχει πει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση το θέμα των ανοιχτών δεδομένων. Γιατί αν τα δεδομένα είναι μια τόσο σημαντική κληρονομιά, δεν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας για τα ανοιχτά δεδομένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χριστόφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η νέα πράσινη συμφωνία ή το νέο πράσινο σύμφωνο θα επιτρέψει ε, στην Ευρώπη να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη βιομηχανία μας. Ενώ ε, οι ανταγωνιστές μας δεν εγκαταλείπουν κατά ανάγκη τους παραδοσιακούς ε, ενεργειακούς τους πόρους. Πώς θα στηρίξετε την ανταγωνιστικότητά μας, πώς θα βοηθήσουμε τη βιομηχανία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσει τη νέα πράσινη συμφωνία. γιατί υπάρχουν και εθνικέ ιδιαιτερότητε. Η πυρηνική ενέργεια σε κάποιε χώρε θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητά του. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκέρ. Ε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Συμφωνώ με του συναδέλφου που ρώτησαν για το ρόλο των παραδοσιακών βιομηχανιών. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή χαλιβουργική στην ε, Γερμανία. Παίζει σημαντικό ρόλο η χαλιβουργία εκεί. Οπότε χρειαζόμαστε, είναι στρατηγική αυτή η βιομηχανία για μα. Είχαμε τεράστια ανάγκη σε επενδύσεις ε, και όπως είπε και ο κύριος Μπούζεκ, ε, ε, μεταξύ άλλων χρειάζεται άνθρακα. και υπάρχει απειλή λόγω των σημερινών συνθήκων μας ανησυχεί ο συνοριακός φόρος άνθρακα και με τα μέτρα που θα ληφθούν ε, ε, με το χάλιβα από χώρες ε, όπου παράγεται χάλιβας χωρίς τέτοια προβλήματα και με ανησυχεί όταν μου λέτε ότι η βιομηχανική πολιτική μας στρατηγική θα αλλάξει υπό αυτή την έννοια. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στον Επίτροπο γιατί πολλοί άριθμες ερωτήσεις υποβλήθησαν και όχι εύκολες. Ε, να δώσω το λόγο με... και μετά στην κυρία Γκρίφιν για ένα λεπτό για να μας αποχαιρετήσει και επισήμω. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ελπίζω να μας ξανάρθετε γιατί βλέπετε είναι πολύ ζωηρό το ενδιαφέρον. Φαντάζομαι δεν έχω ένα λεπτό. Οχτώ, οχτώ λεπτά έχετε. Α, μάλιστα. Αν μη τι άλλο, ήσταν σαφεί. Καταρχήν, σα ευχαριστώ εκ βάθου καρδία για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που θα βοηθήσει ιδιαίτερα ε, να επαναπροσανατολίσω τις προτεραιότητές μας. Δεν πρόκειται περί παρεξήγηση. Είναι ευρύτατο το χαρτοφυλάκιό μου και όλα τα θέματα είναι σημαντικά. Και όταν μιλούμε για τη βιομηχανία, εννοούμε όλου του βιομηχανικού τομεί. Φυσικά και η ψηφιακή επανάσταση θα αλλάξει τα πράγματα. Αλλά στόχο μου είναι το σύνολο τη βιομηχανία και η παραδοσιακή βιομηχανία να παραμείνει και να αναπτυχθεί. Γιατί πάντα θα χρειαζόμαστε και τις παραδοσιακές ε, μορφές βιομηχανίας, τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους και θέλουμε τα εργαλεία για να προσαρμοστεί και η παραδοσιακή βιομηχανία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στόχος μου είναι να την προστατεύσω γιατί θα έχουμε μετάβαση χρονοβόρα και σίγουρα αυτή η μετάβαση εγείρει ανησυχίε που είναι πολύ εύλογες και θεμητές και στόχος μου είναι να ε, προβλέψω τα εργαλεία ώστε να συμπαρασταθώ στην παραδοσιακή βιομηχανία, σε όλους τους κλάδους της. Και επίσης οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε σήμερα θα είναι μακροπρόθεσμες. Θα έχουν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα. Και είπαμε να μην αφήσουμε κανένα στο περιθώριο, να μην αφήσουμε κανένα ουραγό. Αυτό συμφώνησα με τον συνάδελφο Νικόλο Σμιτ. Και η βιομηχανία μας χρειάζεται αυτά τα κρίσιμα υλικά που προέρχονται από κάποιες πηγές ανεφοδιασμού. Τον κατάλογο θα τον προσδιορίσουμε, θα τον ενημερώνουμε, θα τον επικαιροποιούμε και θα ήθελα στην αξιολόγηση των γεωπολιτικών κινδύνων που ε, συνδέονται με τον ανεφοδιασμό μας σε πρώτες ύλε. θα πρέπει να δούμε τι ε, έχουμε στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πολλά χρήσιμα υλικά και κρίσιμα υλικά στην Ευρώπη που δεν έχουμε, α, δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί. Μερικές φορές δεν γνωρίζουμε τι κοιτάσματα έχουμε. Θα αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες με τη νέα γενιά του Κοπέρνικος για να χρησιμοποιήσουμε και τις κβαντικές τεχνολογίες και να γνωρίσουμε καλύτερα το ευρωπαϊκό υπέδαφος, που δεν το γνωρίζουμε ακόμη καλά. Η ενεργειακός έλεγχος, ενεργειακό μείγμα και συμπαράσταση στη βιομηχανία και την παραδοσιακή. Αυτά είναι προτεραιότητες μου. Παρόλο που σήμερα δώσαμε περισσότερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα, γιατί αυτό ήταν το πρώτο θέμα που θα παρουσιάσω και η πρώτη πρωτοβουλία σε αρχές Μαρτίου. Γι' αυτό στάθηκα λίγο περισσότερο σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνώ τα υπόλοιπα. Ή μάλλον αρχές Φεβρουαρίου, όχι Μαρτίου. Και το όραμά μα είναι πολύ πτυχό. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μου είναι προσφυλές, παρόλο που δεν το ανέπτυξε ιδιαίτερο, το θέμα των υπηρεσιών. Ίσως δεν το συζητήσαμε εκτενώς, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει στις συζητήσεις είναι στις βιομηχανικές δραστηριότητες να αναπτύσσουμε και τις υπηρεσίες και για αυτό το θέμα θα έρθω κάποια άλλη στιγμή να σας μιλήσω. Ο κύριος Γκούτλερ μίλησε για την νομοθετική πράξη «Αγοράστε ευρωπαϊκά» by European Act. Δεν μου αρέσουν και πολύ τα σλόγγαν, αλλά όντως για κάποιους τομείς σήμερα θέλουμε περισσότερη κυριαρχία. Μιλήσατε για την άμυνα, ε, διαστημική πολιτική επίσης. Ε, ατομικά ορολόγια. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν κάποια σημαντικές συνιστώσεις. Ήδη υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα διατρανώνουμε και όλα. Πάντως ξέρετε που στέκομαι εγώ σε σχέση με, αυτή την προ... με αυτό το θέμα, αυτό το προβληματισμό. Επίσης, άμεσα ή έμεσα αναφέρεται σε αυτόν τον περίφημο μηχανισμό προσαρμογή του άνθρακα στα σύνορα, του συνοριακού φόρου άνθρακα. Στο μηχανισμό αυτό, πίσω από το μηχανισμό αυτό, υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό που είναι συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού. Και σε αυτή τη φάση του μετασχηματισμού, τη ρηξικέλευτη ε, μετατροπή ε, και του τομέα των υπηρεσιών μα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε θεμητό ανταγωνισμό. Έχουμε μηχανισμού και εργαλεία. Και το είπαμε με τον Φιλ Χόγκαν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς ώστε τα προϊόντα και τα αγαθά που φτάνουν στην Ευρώπη, τα εισαγόμενα προϊόντα και αγαθά, να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές και πρότυπα που πληρούν και τα δικά μας εγχώριας παραγωγής προϊόντα. Αυτό ισχύει για τους κοινωνικούς ε, κανόνες, ε, για τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Δεν είναι μόνο ο συναριακός μηχανισμός του άνθρακα. Αυτό σχετίζεται με το New Green Deal, αλλά υπάρχουν και άλλα εργαλεία και θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο με τον συνάδελφο Χόγκαν για να δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Θα έρθουν και άλλες ε, βιομηχανίες που θα μας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε λοιπόν να μας αποσταθεροποιήσουν σε αυτή τη μεταβατική φάση της βιομηχανίας μας. Σε όλα αυτά τα θέματα αφιερώνουμε ιδιαίτερο χρόνο και προσπάθεια και εγώ και ο Φιλ Χόγκαν. Κάποιος μίλησε για το ρόλο της Ευρώπης που βρίσκεται ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Είμαστε μία ήπειρος με οικονομικό βάρος εφάμιλο για να μην πω ανώτερο των σημαντικών εταίρων μας και των ανταγωνιστών μας. Οπότε μπορούμε να συγκρινόμαστε, αλλά να μην είμαστε και αφελείς. Και όποιες και θα είναι οι επόμενες μας σχέσεις, οι μελλοντικέ μας σχέσεις, γιατί σίγουρα η πολυμέρεια έχει τροποποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, και έχουμε όλο και περισσότερες ανταλλαγές. Αυτές οι ανταλλαγές όμως φαίνεται ότι όλο και περισσότερο θα γίνονται προσπαθώντας να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό από όπου και αν προέρχεται. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σίγουρα ταλανίζεται κάπως από τη γραφειοκρατία της και ο Τραμπ τις προτάσεις του ενισχύει την προεκλογική του εκστρατεία και αναφέρθηκε σε έξι σημεία. Εμεί θα επικεντρωθούμε σε ένα για να δούμε αν θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και σίγουρα αυτός θα είναι σημαντικός στόχος της Επιτροπής μας. Πολύ, ε, πολύς λόγος έγινε και για τη διαστημική πολιτική. Φυσικά, στο διάστημα είναι σημαντικό να είμαστε αξιόπιστος παράγοντας και εταίρος. Και εγώ πρόσφατα μίλησα για το πρόβλημα της διακυβέρνησης που έχουμε με τον Γαλιλαίο. Εξέτασα το θέμα και διαπίστωσα ότι ένα από τα περιστατικά που είχαμε το καλοκαίρι ευτυχώς αφορούσε μόνο κακή διακυβέρνηση γιατί φοβήθηκα μήπως οφειλόταν σε άλλες αιτίες γιατί για μια εβδομάδα περίπου διεκόπη η υπηρεσία και όταν έχουμε ένα δισεκατομμύριο χρήστε, δεν είναι λίγο. Πάντω ήταν ένα θέμα κακού συντονισμού, κακή διακυβέρνηση. Γι' αυτό, σε συνεργασία με του εταίρου μα, θα προτείνω μια νέα διακυβέρνηση που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, γιατί ο κανονισμό δεν εφαρμόστηκε ακόμη. Και θα πρέπει να συν, συντονιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους αρμόδιους φορεί για να καταλήξουμε σε σωστή και βελτιωμένη διακυβέρνηση. Το θέμα της χρηματοδότησης βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αναφερθήκατε και εσείς, το αναφέρατε και εσείς, ε, ισχύει και για το διάστημα και για τα ψηφιακά και για την αμυντική βιομηχανία. Ε, πρόκειται για θέματα τα οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά και για το μέλλον και για την ανθρωπότητα και για την Ευρώπη και επομένως ε, ε, πραγματικά ε, όλα αυτά αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης ε, και ε, χρειαζόμαστε υποστηρίξη έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το επίπεδο το οποίο αρχικά είχαμε ε, θεωρήσει ως στόχο. Όσον αφορά την ε, κυβερνοασφάλεια, βεβαίω συμφωνώ μαζί σας. Από την άλλη μεριά θα μπορούσαμε σε μια μικρή επιτροπή να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Πάντως, σαν γενική αρχή λέω ότι συμμεριζόμαστε απολύτως την προβληματική αυτή 85% των δεδομένων ε, ε, μέχρι το 25 ε, θα αποθηκεύονται παντού και όχι μονάχα στα data centers, στο cloud και επομένως θα αλλάξει τελείως το υπόδειγμα και το αφήγημα της κυβερνοασφάλειας και μέχρι τώρα είχαμε την επιφάνεια επίθεσης κατά κάποιο τρόπο μέσα στα ε, κέντρα, τώρα θα είναι ε, πολύ πιο απλωμένο, θα πρέπει να ξαναδούμε επομένω και να ξαναδουλέψουμε ε, πάνω σε όλα τα στοιχεία. Και βεβαίως ξέρω ότι υπάρχει και από πίσω όλη η συζήτηση για το Cyber Research Center και πρόθεσή μου, σκοπός μου είναι να δουλέψω γρήγορα έτσι ώστε ακόμα και η υποκρατική ε, προεδρία να ληφθεί απόφαση για την υλοποίηση ε, αυτού του κέντρου και ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσά ε, γιατί παίζετε σημαντικό ρόλο. Ε, σε αυτό το θέμα. Ε, βεβαίως η χρηματοδότηση, η, πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και των ε, νεοφυών επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε περισσότερα εργαλεία. Άλλωστε αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μας διαφοροποιεί από τις ΗΠΑ. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στην Ευρώπη. Ωστόσο γίνεται πολλά όσον αφορά τα δεδομένα, πολλές είναι και οι, ε, οι νεοφυείς ε, ε, επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν πάνω στα δεδομένα, οι οποίες χρησιμοποιούν όλα τα στοιχεία της ψηφιακή εποχής, άρα είμαι αισιόδοξο. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, αυτή, αυτός ο συνοριακός ε, φόρος άνθρακα, αυτός δηλαδή προσαρμογής ε, στα σύνορα, δεν θα κάνουμε πίσω. Το λέω και το επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε την ε, μετάβαση. Επομένως, ναι, χρειαζόμαστε και πόρους στην Ευρώπη, άρα είναι καλό να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα μας δίνει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε αυτήν την μακρά μετάβαση. Ε, μιλάμε για δεκαδείς, ε, για την Πράσινη Συμφωνία δεν είναι λίγα χρήματα. Ε, να πω και δύο λόγια σε αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά ε, με τον ε, ε, ελάχιστο αξιοπρεπή μισθό, καθώς επίσης και τη δυνατότητα της 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη και για όλο τον πληθυσμό. Ναι, βεβαίως υπάρχει το θέμα του κόστους των αδειών. Ε, και ε, ναι, πρόκειται για ε, πόρο που θα βρίσκεται στα χέρια των κρατών των κυβερνήσεων. ναι, μίλησα περισσότερο από όσο μου είχατε πει. Encore συνάντησα πριν από λίγο καιρό ε, και στην προετοιμασία της ακροασής μου. Είναι εξαιρετικό ε, που έχω την ε, δυνατότητα να απευθύνομαι και να συζητώ με βουλευτές που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Βεβαίως εγώ έχω υπάρξει υπουργός οικονομικών, έχω πολλές επαφές με το εθνικό μου και εθνικά κοινοβούλια γενικά. Εδώ είναι άλλη διάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που είχα την δυνατότητα να ανταλλάξω από απόψεις ε, ε, μαζί σας για πολλά θέματα. Βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε άλλη φορά και για τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, μπορούμε να μιλήσουμε για τη βαριά βιομηχανία. Βλέπετε ότι τώρα είμαστε πια οργανωμένοι, έχουμε όλες ε, τις ομάδες και μπορούμε να δουλέψουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Μην φύγετε δύο λεπτά ακόμα για να ακούσουμε και τη συναδέλφα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Αναμένουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη με ανυπομονησία και τη δική σας θέση για τη βιομηχανική πολιτική και φυσικά θα μας κάνει μεγάλη τιμή να ξανέρθετε στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε λεπτομερώς του τομείς που αναφέρατε μετά τώρα για τα διάφορα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τερεζαντέθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, οι βουλευτές, οι εργατικοί από τη Βρετανία ήθελαν να παραμείνουν. Είμαστε και Βρετανοί και Ευρωπαίοι. Οπότε προς όλους τους νέους ανθρώπους στην περιοχή μου που ψήφισαν να παραμείνουμε, ζητώ συγγνώμη. Ήθελα να αποτισώ φόρο τιμή, ε, αν με επιτρέπετε, στην κόρη μου Μπρέτα Γκριφίν που τα τελευταία 34 χρόνια μου συμπαραστάθηκε σε αυτό το καταπληκτικό ευρωπαϊκό έργο και ε, έχετε πει σωστά, ήταν πολύ καλό διανοητική διοκτησία, το κλίμα, η ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή ένδυα, η αλληλεία. Ένα σωρό ανθρώπου θέλω να ευχαριστήσω, το προσωπικό ασφαλεία, τα μέλη, τους διερμηνείς, τους συμβούλους, ε, Τζέρεμι, Έμιλι, τον Κρι Πόλς, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε δουλέψει χωρίς εσένα, τον Κρι Βίλιαμ, τη Σάρλοτ, τον Φρέζερ, την Τάρια και πολλού άλλους και τους συναδέλφους μου, τους ευρωβουλευτές που συνεργάστηκαν μαζί μας για το δέσμε μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι εδώ βοηθάμε τους ανθρώπους. Πέτρα Ματσίνα, Μαρία Εντουάρντ, Εσμελ, Σολεντάντ, Ντάν, Κάρλος, Κορνίλια, Μίριαμ, Γιούτον, Κριστιαν, στο ΣΕΝΚΟ που μου έδωσε αυτό το παραπάνω μισό της εκατό για την ενεργειακή απόδοση. Και για την ενεργειακή απόδοση θα ήθελα να πω για όλους, για κάθε 1% αύξηση στην ενεργειακή απόδοση. Γίνεται δυνατή ανακαίνιση 3 εκατομμυρίων σπιτιών και 7 ε, εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν από την ενεργειακή ένδυα στην Μισελ Ραβεσί στον απερίγραπτα καλό Κλοντ Τέρμες και Μπιουζέκ ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ αλλά σταμάτα να πατάς τόσο πολύ τον γκάζι. Το Μιγγέλ μας, το Κάρλος, τους επιτρόπους μας, τους νέους βουλευτές μου, τους Γιάννη, στον συνάδελφό μου που βρίσκεται δίπλα μου, στους νέους επιτρόπους, στο προσωπικό, στη Λόρα, στον Αντώνιο που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα. Αλλά αν με επιτρέπετε, ήθελα να κλείσω με ένα τραγούδι από το Λίβερπουλ, το οποίο έχει ως εξής. Όταν περπατάς με στην καταιγίδα, κράτα το κεφάλι σου ψηλά και μη φοβάσαι το σκοτάδι. Αφού περάσει η καταιγίδα, σε περιμένει ένας χρυσός ουρανός. Ένα γλυκό, ασημένιο τραγούδι, τύχης. Περπάτα μέσα στον άνεμο, συνέχισε να περπατάς μέσα στη βροχή, παρότι τα όνειρά σου έχουν χαθεί. Συνέχισε να περπατάς, συνέχισε να περπατάς με ελπίδα μέσα στην καρδιά σου και ποτέ σου δεν θα βρεθείς να περπατάς μόνος. Η Βρετανία είναι μαζί σας. Δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς και όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκατε στην Επιτροπή Ήτρα μέσα στα χρόνια. Σας αποχαιρετούμε και ελπίζουμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή και κοντά στο μέλλον. Colleagues, we see each Θα τα πούμε στις 17 Φεβρουαρίου, αγαπητοί συνάδελφοι.